Ε, στις 22 Οκτωβρίου ε, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη και σας προτείνω εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων να γίνουν εξής αλλαγές στην τελική ημερήσια διάταξη. Οι δύο δηλώσεις της Αντιπροέδρου της ε, ΥΠΑ της εκπρόσωπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής για την κατάσταση του Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και την κατάσταση του Νότιου Σουδάν θα μεταφερθούν από την Τετάρτη το απόγευμα στην Τρίτη το απόγευμα μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η δήλωση τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 καθώς και η έκθεση όρου θα μετάφερθουν από Τετάρτη απόγευμα σε... από Τρίτη απόγευμα σε Τετάρτη απόγευμα πριν την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μάλιστα. Άρα εγκρίνονται έτσι οι αλλαγές στην ημερήσια διατάξη. Έχετε το λόγο κύριε Ρούμπιχ. Μία έκκληση. Η ψηφοφορία το, την Πέμπτη. Οι ψηφοφορίες θα είναι ε, πάρα πολύ μεγάλες και ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μισή ώρα πιο νωρίς. Ναι, κοιτάξτε, μόλις φτάσουμε στην Πέμπτη, λέει ο Πρόεδρος. Έχει γίνει ήδη αυτή η αλλαγή που ζητάτε δεν είχε να κάνει με την αλλαγή της ώρας. Είχε να κάνει με την ε, πιο πρωινή κίνηση των ψηφοφοριών. Το, η ομάδα του ΕΛΚ με δήλωση, ζήτησε μάλλον δήλωση της είπα εκπροσώπου για την γεωργία και ιδιαίτερα για την κατάσταση του τηλεοπτικού σταθμού Ρουστάφη 2. Ζήτησε λοιπόν να μπει αυτό για την Τετάρτη το απόγευμα με ψήφισμα. Υπέρ του αιτήματο δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω παρά τα θέματα που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων ε, να κοιτάξουμε στη μήνυ ολομέλεια μάλλον σε, να μην μπουν στη μήνυ ολομέλεια, αλλά τώρα να μπουν τα θέματα αυτά. Γιατί τώρα θα ληφθούν οι αποφάσεις για αυτή την υπόθεση. Γιατί αν είναι να τα αποφασίσουμε αυτά και να κάνουμε ε, το ψήφισμα στη μήνυ ολομέλεια, θα είναι μόνο για να ε, υποβάλουμε ένσταση κατά μια απόφαση. Τώρα μπορούμε να αποτρέψουμε και μια απόφαση και δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια τη Ανατολική Συντηρική σχέση με μια χώρα που έχουμε συμφωνία σύνδεση. να μπορούν να παραλύσουν η κυβέρνηση την τελευταία, τον τελευταίο τηλεπτικό σταθμό που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι είναι θέμα αρχής, θέμα ελευθερίας έκφρασης. Ξέρω ότι υπήρχε ζήτημα για να μπει στο Νοέμβριο, στην Ολομέλεια του, Νοεμβρίου το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρας δεν έχω ζητήσει ποτέ πραγματικά τίποτα στα πλαίσια αυτή του καταπήγοντο χαρακτήρα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπρόκ, λέει ο Πρόεδρο. Ποιο θα ήθελε να υποστηρίξει το αίτημα του κύριου Μπρόκ. Υπέρ, λοιπόν. Κανεί. Ποιο είναι κατά. Η κυρία Χάουταλα. Um, Πρόεδρε, θέλω να απευθύνω έκκληση προς όλους μας να μην μπει το θέμα αυτό στην μέση διαταξή αυτή την εβδομάδα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αντιπροσωπεία θα μεταβεί εκεί στο τέλος της εβδομάδας και θα είναι η πρώτη συνάντηση με την Γεωργία ιστορικά και θα ήταν κρίμα να λάβουμε θέση τώρα. Βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τους συναδέλφους και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση το θέμα αυτό στην επίσκεψή μας στη Γεωργία. Να τονίσω επίσης ότι όταν είχε τεθεί αντίστοιχη περίπτωση με την προηγενέστερη κυβέρνηση το κλείσιμο της τηλεόραση του τηλεοπτικού σταθμού η Μέντι από την κυβέρνηση δεν υπήρξε αντίδραση από αυτούς που τώρα θέλουν να προτείνουν ψήφισμα. Τρίτον, ως συμπρόεδρος της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest ανησυχώ πολύ διότι φοβούμαι ότι βλάπτουμε την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου με διπλά επίπεδα, με, με διαφορετικά στάνταρ. Δεν μπορεί να μην έχουμε την ίδια στάση σε όλους τους εταίρους στην Ανατολική Ευρώπη. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα για το αίτημα η κατάσταση στη Γεωργία και η κατάσταση του σταθμού Ρουστάβε 2. Το αίτημα λοιπόν είναι να μπει σε αυτή την ολομέλεια το θέμα αυτό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. Αλλά Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Die Abstimmung Πέρας σου. Απορρίπτεται. Και παραμένει λοιπόν απαραλλαχτή μερίσια διάταξη. Κυρίε και κύριοι, η Ενωμένη Αριστερά, η Γκουε, ζητά δήλωση τη είπα τη ε, εκπροσώπου για την 40η ε, επέτειο του πράσινου Μάρτη στην Δυτική Σαχάρα, την Τετάρτη. Η κυρία Σάντσες η κυρια Σάντσο καλντενα θα πάρει το λόγο για να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 6 Νοεμβρίου έχουμε τα 40 χρόνια από την πράσινη πορεία και κατοχή ε, της Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο. Ε, έδαφος που έπρεπε να, να αποαπικιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 73 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσέχει την πολιτικά τη σύγκρουση αυτή και συμβάλλει στην ε, παγίωση του status quo διατηρώντας σε παράλυση τα σχέδια των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή αυτή. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να υπερασπίζεται τα, δι... τα δικαιώματα του ανθρώπου όπως διατείνεται, αυτό το θέμα πρέπει να μπει επιτάπητος. 90.000 άτομα και βρίσκονται εδώ και 40 χρόνια εκτός της χώρας τους λόγω της κατοχής από το Μαρόκο. Πρόσφατα ε, βροχ, τεράστιες βροχές κατέστρεψαν την περιοχή του Ντιντούφ όπου είναι τα στρατόπεδα των προσφύγων. Ζητώ την υποστήριξή σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφα. Ποιος θα ήθελε να υποστηρίξει το αίτημα της συναδέλφου. Κύριε Λάμπερτς, έχετε το λόγο. Δεν μιλώ, δεν παρεμβαίνω γιατί πρόκειται για μια πράσινη επέτειο. Η επέτειος αυτή θα έπρεπε να γίνει και στην μήνυ ολομέλεια του Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, άρα μπορούμε να δεχθούμε το αίτημα της ομάδας Γκουε κάνοντας τη συζήτηση αυτή στην σύνοδό μας στη ε, συνεδρίαση της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, αλλά είναι για άλλο αίτημα που πήρατε το λόγο. Ναι, μεν μιλήσατε για το περιεχόμενο και υποστηρίξατε το περιεχόμενο του αιτήματο, αλλά δεν υποστηρίξατε το ίδιο το αίτημα. Ποιο θα θέλει να πάρει το λόγο κατά του αιτήματο τη κυρία Σάντσοε, κύριε Πρέντα. Ε, ε, Πρόεδρε, φοβάμαι καταρχά ότι είναι κάπω ε, πρόημο να συζητήσουμε για τι 6 Νοεμβρίου Οκτώβριο είμαστε. Ξέρω ότι οι κομμουνιστές ε, τις επαιτίους ε, τις ε, γιορτάζουν νωρίς. Αλλά δεν πρέπει να πάμε τρέχοντας. Επίσης δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εδώ. Ξέρω ότι είναι σημαντικό ζήτημα που συζητείται στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Δεν νομίζω ωστόσο ότι είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν βλέπω ε, το λόγο. Αν γίνει μια ανταλλαγή απόψεων στην αντιπροσωπεία του Μαγκρέμπ, ίσως, αλλά πρώτα πρέπει το αίτημα να έρθει από την ε, ομάδα, από την Επιτροπή για το Μαγκρέμπ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ο συνάδελφος Λάμπερς είπε ότι θα μπορούσαμε να διαβουλευτούμε και τον Νοέμβριο. Αποσύρετε λοιπόν το αίτημά σα Και η ομάδα ζητά να μπει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου και θα μπει στο σχέδιο της μέρης της διάταξης. Ε, υποστηρίζουμε την πρόταση Λάμπερς να περάσει στη μήνυ Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Μάλιστα λοιπόν, ούτε θα βράξουμε. Και τώρα θα ήθελα να σας ε, ζητήσω στην προπαρασκευαστή συνάντηση, κυρία Τσίμερ, ε, τη διάσκεψη των Προέδρων να το συζητήσουμε αυτό και να δούμε κατά πόσο θα μπει ή όχι στην ημερήσια διάταξη. Και έτσι λοιπόν δεν επηρεάζεται η ημερησία διάταξη για την εβδομάδα αυτά. Ο συνάδελφος Ρούμπιχη για την Πέμπτη ζήτησε να ξεκινήσουμε πιο νωρίς κατά 30 ή 45 λεπτά τις ψηφοφορίες. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος του κ. Ρούμπιχη. Όχι, δεν είπα να ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, χαίρομαι που είσαστε όλοι υπέρ, αλλά είναι κανείς κατά. Είναι κανείς κατά του αιτήματο. Ζητώ λοιπόν επίσημα ποιος θέλει να ξεκινήσουμε πιο νωρί τι ψηφορίε 30 έω 45 λεπτά. Κατά. Αποχές. Πρώτη φορά εδώ στο Κοινοβούλιο ομόφωνη απόφαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο πράγματα θα ήθελα να σας επισημάνω ωστόσο. Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν 30 λεπτά πιο νωρίς. Αυτό μειώνει το χρόνο αγόρευση των ομάδων κατά 30 λεπτά. Και όλους όσοι διαμαρτυρηθούν που έχουν λιγότερο χρόνο αγόρευση, θα στείλω το, τα email τους ε, σε αυτούς που πήραν την αποφάση σήμερα. Κύριε Καστάλτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να υπογραμμίσω το εξή. Συχνά την Πέμπτη το πρωί βρισκόμαστε να συζητάμε τα κατεπήγοντα, όπω και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ε, περικοπή πάνω από μισή ώρα του χρόνου που θα έχουμε στη θέση μου. Συμμερίζομαι το αίτημα του κυρίου Ρούμπιχα, ε, όμω υπογραμμίζω ότι πολύ συχνά τα κατεπήγοντα δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, τόσο επειδή λείπουν πολλοί συνάδελφοι, όσο και επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να το συζητήσουμε. Δεν θα ήταν καλύτερο να μετακινηθούν όλα τα κατεπήγοντα για τις ολομέλειες των Βρυξελών. Διατυπώνω αυτό το αίτημα και ελπίζω πως το Προεδρείο θα το λάβει υπόψη και θα το σκεφτεί. Κύριε Καθάλτο, καταλαβαίνω απόλυτα το αίτημά σα, αλλά δυστυχώ θα πρέπει να σα ενημερώσω ότι την Τετάρτη δεν έχουμε καθόλου. Την Πέμπτη, μάλλον, δεν έχουμε λέει κανένα. Ε, κατεπήγον στην μερική ο Πρόεδρο. Μόνο κανονικέ συζητήσει. Και επειδή τον Οκτώβριο έχουμε πάντα δύο ολομέλειες, στη δεύτερη ολομέλεια δεν έχουμε κατεπήγοντα, αλλά το συμπεριλαμβάνουμε για την επόμενη φορά. Και έχουμε και την πέμπτη το απόγευμα ως ημέρα εργασίας επιπλέον. Κυρίε και κύριοι, τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης στη συζήτηση για τα θέματα της φορολογίας. Και καταρχάς έχουμε την έκθεση Φέρμπερ για την υποχρεωτική ανταυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. να διευκρινίσω κάτι και να απαντήσω για το θέμα της έλλειψης ε, χρόνου και τη δυνατότητα μετακίνησης των συζητήσεων στη μήνυ ολομέλεια των Βρυξελών. Εγώ θέλω να παρέμβω για να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που ήδη προβλέπεται για την συνεδρίασή μας εδώ στο Στρασβούργο. Θυμίζω ότι πέμπτη απόγευμα είναι χρόνος ολομέλειας. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την πέμπτη απόγευμα όπως προβλέπεται από τις συνθήκες ούτω ώστε κατόπιν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μεταφέρουμε και άλλες συζητήσεις κατόπιν της Βεξέλλης. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, δεν ακούσατε ίσως αυτό που είπα. Δεν με ακούτε, ούτε τώρα. Κύριε Ζάντερ, εδώ και ένα λεπτό προσπαθώ να απευθυνθώ προς εσάς, αλλά δεν με ακούτε. Αυτό ακριβώς είπα, ότι έχουμε και την πέμπτη απόγευμα, ως μέρα δουλειάς. Βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος.